η προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή 20, του κανονισμού 2157-2001 του Συμβουλίου της 8 Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Με πρώτον ο ε, ομιλητή τον κύριο Λένε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, <clears throat> περί τίνος πρόκειται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2001 έλαβε μια απόφαση σχετικά με το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεφαλουχικής Εταιρείας. το οποίο όμως τέθηκε για ρεφόρους λόγους σε ισχύ την 1η 8 2004. Και όπως συμβαίνει συχνά, παρακαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την πάροδο κάποια ε, περίοδου να συντάξει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία και από αυτή την έκθεση να μπορέσουν να συναχθούν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη ενδεχομένω να γίνουν κάποιε τροποποιήσει. Αυτό, όπω είπα, τον Οκτώβριο του 2004, Οκτώβριο, αύριο λοιπόν είναι λίγη προθεσμία των πέντε ετών. Δεν υπάρχει όμως έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή όλοι τηρούμε τον νόμο και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεματοφύλακα των συνθήκων καλείται να τηρεί επίσης τους ευρωπαϊκούς νόμους, εμείς στην Νομική Επιτροπή αποφασίσαμε να ερωτήσουμε τι γίνεται. Για ποιο λόγο δεν έχει ακόμη υποβληθεί η σχετική έκθεση, ούτε έχει συνταχθεί. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεμελιώσει την στάση της να καταστεί σαφέ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι δύο Συνομική Επιτροπή ασκούν το ελεγκτικό του καθήκον απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα εξατλήσω τα πέντε λεπτά που μου έχετε διαθέσει. Θα χαρώ ιδιαίτερα εάν μπορέσει ο κύριο Επίτροπο, μετά από αυτή την σύντομη προφορική μου εισαγωγή να απαντήσει. Η πρόεδρο. Σα ευχαριστώ κύριε Λένε. Κύριε Ταγιάννη, εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω εξ ονόματο του Επιτρόπου Μακρύβη, τον οποίο αντικαθιστώ σήμερα, την Νομική Επιτροπή, τον Πρόεδρο Λένε, που έθεσαν αυτό το θέμα. Μιλάω εξ ονόματο του Επιτρόπου Μακρύβη. Και χαίρομαι που το Κοινοβούλιο ασκεί τον ελεγκτικό του ρόλο. Γιατί νομίζω ότι οθεί την Κομισιόν να δουλεύει καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τα δύο πρώτα ερωτήματα τα οποία ετέθηκαν, με χαρά σας ενημερώνω ότι οι εργασίες για την προετοιμασία της έκθεσης ε, ε, έχουν προχωρήσει πολύ. Η Κομισιόν ζήτησε μία μελέτη εξωτερική που θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του 2009 και θα αποτελέσει αυτό μία βάση για την εκπόνηση της έκθεσης. Η Κομισιόν θα αναλύσει με, εμβαθή, με ενδελεχή τρόπο αυτή τη μελέτη και θα ακούσει με προσοχή τον την άποψη των ενδιαφερομένων. Η έκθεση λοιπόν θα δημοσιοποιηθεί το δεύτερο εξάμεινο του 2010 και θα διαβιβαστεί και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Φυσικά, οι προθεσμίες θα αποφασιστούν από την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση θα αναλύσει τις τέσσερις δυνατότητες τροποποίησης που προβλέπονται ρητός από το άρθρο 69 του κανονισμού και σε αυτή τη φάση η Κομισιόν δεν έχει ακόμα θέση για τις πιθανές τροπολογίες ε, του καταστατικού. Θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της εξωτερικής μελέτης και της διαβουλεύσης. Θα πρέπει να ελέγξουμε κάθε παράγοντα ε, και τις ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για το καταστατικό της ε, Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Και φτάνω τώρα στο τρίτο ερώτημα. Οι, χρόνοι που... και οι προθεσμίες που θα προβλεφθούν. Αυτές θα αποφασιστούν από τη νέα Επιτροπή. Και είμαι πεπισμένος ότι θα προσέξει πάρα πολύ αυτό το θέμα και φυσικά θα ακούσει και την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν υιοθετήσει ε, ενδεχόμενα μέτρα ή ενδεχόμενα νομοθετικά κείμενα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η ενδεχομενα νομοθετικα κειμενα σας ευχαριστω λεει Η επόμενη αγορήτριά μας είναι Απούσα. Προχωρώ στους υπολείπους συναδέλφους που έχουν ήδη εγγραφεί. Ο κ. Κούτας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η ιδέα αυτή της Ευρωπαϊκής Εταιρείας έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του 50 και αφού ξεκίνησε δηλαδή η συνθήκη της Ρώμης υπέρ της ε, κοινή αγοράς. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχει μια συμβολική αξία. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή επιχείρηση η οποία χαίρει κάποιας ελευθερίας εγκατάστασης και κάποιας κινητικότητας. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το καταστατικό αυτό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας. Πρόκειται για ένα μέσο που έχουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν την διασυνοριακή τους προσπάθεια συγχωνεύσεως. Αυτό είναι και ένα από τα πλεονεκτήματα εξάλλου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας ότι η έδρα της μπορεί να μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος εκεί όπου έχει καταχωρηθεί δηλαδή η επιχείρηση σε κάποια άλλη χώρα μέλος χωρίς να χρειάζεται γι' αυτό να δημιουργήσει μια νέα εταιρεία. Παρ' όλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Εταιρεία δεν έχει ένα αυτόνομο καταστατικό που να διέπεται από ενιαία νομοθεσία. Άρα στην πράξη υπάρχουν δυσκολίες. Το καταστατικό συνεπώ δεν είναι ομοιόμορφο και εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία κάθε φορά. Άρα και η κινητικότητα που λέμε τη ευρωπαϊκή εταιρεία περιορίζεται ουσιαστικά από το ένα ή το άλλο κράτος, ανάλογα με το που βρίσκεται. Να λοιπόν, πώς τελικά περιορίζουμε την ελευθερία διακίνησης των εταιριών. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος, πρέπει να συμπεριλαμβάνει μελέτη για την δυνατότητα να υπάρχει έδρα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας συγχρόνως σε διαφορετικές χώρες. Και η έκθεση αυτή πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αναθεώρηση του κανονισμού, ώστε να προχωρήσουμε προς τη δημιουργία ενός αυτόνομου καταστατικού για τέτοιες εταιρείες. δεν επιθυμεί κανείς συνάδελφος να λάβει το λόγο στα πλαίσια της διαδικασία και Δίνω το λόγο στον κύριο Ταγιάννη. Ευχαριστώ ξανά κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρέμβαση του Προέδρου Λένε και των άλλων βουλευτών που συμμετείχαν στη συζήτηση. Φυσικά ο κανονισμός για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας συμπληρώνεται από μια οδηγία σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους. Και ο χρόνος για την εφαρμογή της είναι, ήταν η 8η Οκτωβρίου του 2004. Ε, αλλά δεν υιοθέτησαν όλοι τα απαραίτητα μέτρα εμπρόθεσμα. Ε, μόνο στις αρχές του 2006 συμπληρώθηκε η διαδικασία ε, λήψης μέτρων. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να δούμε αν ο κανονισμός ε, ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ε, για αρκετό χρόνο για να, κάνουμε, να εκπονήσουμε μια έκθεση για την εφαρμογή του. Ε, Επομένω, υπάρχουν καθυστερήσεις και συμφωνώ με τα όσα είπε ο πρόεδρο λένε. Ελπίζω να μπορέσουμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να δώσουμε συγκεκριμένε απαντήσει απαντήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα τη Ευρωπαϊκή εταιρεία. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ε, το δεύτερο εξάμεινο του 2010. Θα απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα, όχι μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έληξε η συζήτηση. Διακόπτεται και η συνεδρίαση. Θα συνεχιστεί αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Σας εύχομαι καλή νύχτα.